Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως την ε, προηγούμενη πέμπτη η βουλευτής Εβίτα Γκριγκούλ με ενημέρωσε πως ε, εγκαταλείπει την ομάδα του EFDD. Την ίδια ημέρα ενημέρωσε την διάσκεψη των Προέδρων πως πλέον το EFDD δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του κανονισμού για το σχηματισμό κοινοβουλευτικής ομάδας καθώς δεν έχει πλέον βουλευτές από 7 χώρες και άρα έχασε το καθεστώς της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παρακαλώ κύριε Βουλευτά. Κύριε Πρόεδρε, αλλάξαμε ή μάλλον αλλάξατε τις θέσεις εδώ αλλά θα ήθελα να πω ότι σήμερα μαζέψαμε τις απαραίτητες υπογραφές ώστε το FTD να παραμείνει ακέραιο. Την περασμένη εβδομάδα παρετήθηκε μία βουλευτής και υποστήκαμε μία πολύ περίεργη επίθεση την οποία βοηθήσατε κι εσείς νομίζω αν δεν την υποδαβλήσατε κιόλας. Ενώ εσείς ως πρόεδρος πρέπει να παραμένετε ουδέτερος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να μας υποσχεθείτε ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια καραγκιοσλίκια στο μέλλον και ότι θα παραμείνετε ουδέτερος όπως προβλέπει, προβλέπουν τα καθήκοντά σας. Κοιτάξτε, οι κοινοβουλευτικές ομάδες σχηματίζονται με βάση τα όσα προβλέπει ο κανονισμό. Άρθρο 32, εκεί πέρα αναφέρεται πω σχηματίζονται οι ομάδε. Όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι βουλευτές από τουλάχιστον 7 χώρες, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου απλά διαπιστώνει δεν έκανα τίποτα παραπάνω ενώπιον της διάσκεψης των Προέδρων. Δεν έχετε πλέον το καθεστώς της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προβλέπονται τα πράγματα από τον κανονισμό. Βουλευτές από 7 χώρες τουλάχιστον που πρέπει να υπογράψουν και να δηλώσουν πως ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Όταν γίνει αυτό θα μου το κοινοποιήσετε και οπωσδήποτε μετά θα κινήσω τις ανάλογες διαδικασίες. Με βάση λοιπόν τον κανονισμό κινήθηκα γι' αυτό και άλλαξε η τοποθέτησή σας εντός της αίθουσας. Και το που κάθονται οι ομάδες ορίζεται στον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά τώρα της ε, συνεδρίας 18 Σεπτεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, ωραία, εγκρίνονται. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Ιζαμπέλα Λεβίν από 3 Οκτωβρίου ε, ορίστηκε Υπουργός Ανάπτυξης της Σουηδίας και την